We will start... Συνάδελφοι, δεύτερο, δεύτερος γύρος ομιλητών της Επιτροπής μας, τάξε 3. Καλωσορίζω τους ε, επισκέπτες μας και το κοινό και τους συναδέλφους. Δεύτερος γύρος ομιλιών. Η ακρόαση θα ασχοληθεί με τα κύρια θέματα και τις προκλήσεις για να αντιμετωπίσουμε τις απάτες του ΦΠΑ. Πρώτα ακούσουμε τον κύριο Νέμπεν Μάτες, που είναι μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου, που θα ασχοληθεί με το θέμα του εάν αντιμετωπίζουμε την ενδοενωσιακή δαπάνη, ε, απάτη. Κατόπιν η κυρία Μάιτε Φάμπρεγα, που είναι στην DG Taxe της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα μας μιλήσει για το τέλος του προσωρινού καθεστώτος και για την απάτη του ΦΠΑ ιδιαίτερα την κυκλική. Κατόπιν η κυρία Άλμα Ντότυρ, από την ε, Σουηδική Εφορία και πρόεδρος του δικτύου Eurofisk. Θα μας μιλήσει για τη συνεργασία των κρατών μελών και τη βελτίωσή της, για την καταπολέμηση της απάτης Καρουσέλ και ποιος είναι ο ρόλος του Eurofisk. Και τελευταίος ομιλητής θα είναι ο κύριος Richard Murphy, ο οποίος είναι στην εταιρεία για φορολογικές μελέτες, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις ενδεχόμενες λύσεις για το πρόβλημα αυτό. Ο κύριος Νέβες Μάτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής, κυρίε και κύριοι. Ευχαριστώ που δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τα κύρια πορίσματα της έκθεσής μας για το θέμα της απάτης του ΦΠΑ και τις επόμενες εκθεσίες μας για τις διαδικασίες αγωγών. Έδωσα αναλυτικές ε, απαντήσεις σε ερωτήσεις σας, οπότε απλώς θα παρουσιάσω μερικά σημεία. είναι, ποια είναι τα κύρια αίτια της ε, απάτης ΦΠΑ. Έχει να κάνει με την ε, τελωνιακή διαδικασία 42 και τις εισαγωγές. Θέλουμε να υπάρχει αυτόματη ένταξη των τελωνιακών στοιχείων στο σύστημα VIES, το σύστημα ανταλλαγή πληροφοριών για τον ΦΠΑ. Το δέχτηκε αυτό η Επιτροπή και το έβαλε στις τροποποιήσεις της οδηγίας για την διοικητική συνεργασία. Ε, έμαθα ότι εγκρίθηκε από το Συμβούλιο, δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη. Αυτό θα διευκολύνει τα στοιχεία από τις ε, διασαφήσεις να μπαίνουν ε, στο VIS και έτσι να μπαίνουν και στις φορολογικές δηλώσεις των εισαγωγέων. Αυτά τα στοιχεία, αυτή η νέα διαδικασία θα ισχύσει την 1η του 2020. Δημιουργήσαμε λοιπόν το νομικό πλαίσιο, αλλά η, στην πράξη εφαρμογή του ακόμη εκκρεμεί. Πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοστεί όσο καλύτερα και όσο ταχύτερα γίνεται αυτός, αυτή η νέα οδηγία. Πού χρειάζεται περισσότερη βελτίωση για την καταπολέμηση της απάτης του ΦΠΑ. Καλύτερη συνεργασία χρειάζεται μεταξύ των ε, φορολογικών αρχών των διαφόρων κρατών μελών. Χαιρόμαστε που η Επιτροπή δέχθηκε τη σύστασή μας να γίνουν περισσότερες ε, επισκέψεις επιτήρησης με βάση την εκτίμηση κινδύνου στα κράτη-μέλη. Το 2017 πήγε σε 10 κράτη-μέλη για την προετοιμασία της έκθεσης για την ε, συλλογή του ΦΠΑ και τις διαδικασίες ελέγχου. Μετά τις επισκέψεις, η Επιτροπή, στα πορίσματά της, έκανε διάφορες συστάσεις σε μια έκθεση για τα κράτη-μέλη για να γίνει πιο αξιόπιστο το VIES, όπως είχαμε ζητήσει και εμείς στη δική μας έκθεση. και ανέφερα στις γραπτές μου απαντήσεις που, συμφωνώ περισσότερο, που συμφωνούμε περισσότερο με την Κομισιόν. Κυρίως όμως πρέπει να υπάρχει καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διοικητικών, δικαστικών και διοκτικών αρχών των κρατών της Ένωσης. Η απάτη του ΦΠΑ είναι από την ουσία του διεθνής, διεθνές εγχείρημα. Ε, οι φορολογικές αρχές ενό ε, κράτου μέλου δύσκολα μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά. Ακόμη και η διμερή συνεργασία δεν επαρκεί. Γιατί τα προϊόντα μετακινούνται μεταξύ διαφόρων χωρών. Στις περιπτώσεις όπου γίνεται μεγάλης έκτασης ε, απάτη. Οπότε θα έπρεπε να παίξουν ε, περισσότερο ρόλο οι ενωσιακές αρχές. Χαιρόμαστε λοιπόν που οι νέες προτάσεις για τη διοικητική συνεργασία που βασίζεται και στις δικές μας συστάσεις από την ειδική έκθεση, προτείνει οι αρμόδιοι του Eurofisk να στέλνουν στοιχεία στη Europol και την Olaf. Και υπάρχει και μια άλλη νέα οδηγία, η οδηγία για τον, τους δημόσιους εισαγγελείς, για τους εισαγγελείς που βελτιώνει τη συνεργασία. Πρέπει επίσης να βελτιωθούν και οι στατιστικές για τις ε, υποθέσεις όπου έχουμε διαπιστώσει τέτοια απάτη. Δεν υπάρχει καμία συστηματική προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Οι προτάσεις τους είναι οι λεγόμενες από πάνω προς τα κάτω εκτιμήσεις για τους φόρους που δεν έχουν συλλεγεί και δεν έχουν ταυτοποιηθεί μάλιστα, αλλά υπάρχουν προβλήματα. Το θέμα είναι πώς ε, θα εκτιμήσουμε το μέγεθος της παραοικονομίας στα διάφορα κράτη-μέλη από την ίδια της τη φύση βέβαια της παραοικονομίας είναι δύσκολο να την εκτιμήσεις. Και η έκταση της παραοικονομίας παίζει μεγάλο ρόλο στην εκτίμηση των διαστάσεων της απάτης. Γι' αυτό πρέπει να βασιστούμε σε υποθέσεις όπου έχει ταυτοποιηθεί τέτοια απάτη. Όπου οι χώρες επιχείρησαν να κάνουν κάποιες τέτοιες εκτιμήσεις. Οι διαφορέ αν η προσέγγιση είναι από πάνω προς τα κάτω ή αντίστροφα, είναι ουσιώδει. Έω και 100%. Καλούμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει κάτι για να συλλέγονται με πιο ε, συγκρίσιμη βάση αυτά τα στοιχεία. Μόνο το Βέλγιο νομίζω και το Ηνωμένο Βασίλειο δημοσιεύουν περιοδικά τέτοια στοιχεία. Θα ήταν ε, σωστό να αξιοποιήσουμε την πείρα αυτών των χωρών για να υπάρξει μια κοινή προσέγγιση σε ενωσιακό επίπεδο. Τέλος. Θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη ανταλλαγή στοιχείων. Τα ε, στοιχεία. Υποτίθεται ότι είναι ε, αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης ε, τα τελωνία. Αλλά επειδή τα κράτη-μέλη ε, κρατούν, το 20% για τα διοικητικά τους έξοδα, είναι περισσότερο μοιρασμένη η αρμοδιότητα. Και αυτό δημιουργεί κάθε είδους αντικίνητρα για να γίνει σωστή συνεργασία. Αν είσαι σε μια χώρα αν είσαι μια χώρα που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εφορίες λένε εάν χάνουμε 100 αλλά το κόστος ε, ε, εντοπισμού αυτού που χάνουμε είναι 50 τότε φυσικά θα επιχειρήσουν να εντοπίσουν ε, την απώλεια αλλά εάν ε, το κόστος εντοπισμού των απολειών είναι μεγαλύτερο από το όφελος, τότε φυσικά δεν θα το κάνουν. Άρα δεν υπάρχει επαρκές κίνητρο για τις αρχές ε, να κάνουν κάτι γι' αυτό. Το άλλο πρόβλημα είναι ότι αυτή η παρακράτηση του 20% των τελωνιακών ε, δασμών και τελών σημαίνει ότι έχεις κίνητρο να υπάρχουν εμπορικές ροές προς τη χώρα σου. Υπάρχουν και άλλα κίνητρα, αλλά και αυτό είναι ένα συμπληρωματικό κίνητρο. Και η έκθεση που ήδη ανέφερα, απεκάλυψε, είναι ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ των χαμηλών εκτιμήσεων που γίνονται για τις απάτες και των εμπορικών ροών προς κάποια σημεία εισόδου. Άρα το σύστημα δημιουργεί κίνητρα για να μην γίνει σωστά η αποτίμηση των απολειών. Όπως είπα, ε, εάν ε, το κόστος για τη συλλογή ενός φόρου είναι 20% του ίδιου του τέλους, είναι πολύ ψηλό. Αυτό το 20% λοιπόν δημιουργεί προβλήματα. Η Κομισιόν τώρα προτείνει να μειωθεί αυτό το ποσοστό παρακράτησης. Αλλά δεν θα λύσει το πρόβλημα. Μπορεί να μειώσει τις διαστάσεις του, αλλά δεν θα το επιλύσει. Γιατί... Θα σας πω την προσωπική μου άποψη, γιατί ως ε, συνέδριο δεν έχουμε πάρει θέση. Αν θέλεις να λύσεις το θέμα αυτό, θα πρέπει να υπάρχει ε, σωστός συνδυασμός του κόστους και ωφέλους. Η πρόταση της Κομισιόν λέει ότι θα πρέπει να μειωθεί 10% η, η παρακράτηση, αλλά θα ε, αντισταθμιστεί με ε, επενδύσεις στις τελωνειακές υποδομές από την Ένωση. Αυτά ευχαριστώ και να απαντήσω στις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μάτες από το ελεκτικό συνέδριο. Η κυρία Μάιτε Φάβρικας Φερνάνδης. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι πολύ που έχω την ευκαιρία σήμερα να σας παρουσιάσω τις απόψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ειδικό αυτό θέμα της απάτης με το ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και να σας παρουσιάσω ε, τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής ε, ε, αγοράς για να δημιουργήσουμε ένα νέο χώρο χωρίς απάτη. Είναι σημαντική πηγή εσόδων ο ΦΠΑ για τους κρατικούς προπολογισμού, αλλά και για τους ιδίους πόρους της Ένωσης. Το 2016 στα 28 κράτη-μέλη τα έσοδα από το ΦΠΑ ήταν περίπου 1,443 ευρώ που αντιστοιχεί στο 18% των φορολογικών εσόδων των κρατών μέλων. Ωστόσο, κάθε χρόνο χάνονται λόγω απάτης μεγάλα ποσά για αποφύπια που δεν αποδίδεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία μας, το 2015 ήταν 151 δισεκατομμύρια ευρώ οι απώλειες που είναι πάνω από 12% των συνολικών αναμενωμένων εσόδων από το ΦΠΑ. Παρόλο που οφείλεται και σε άλλους λόγους αυτό, εκτός από τη φορολογική απάτη. Υπάρχουν πτωχεύσεις ε, και λάθη στους υπολογισμούς, αλλά η απάτη στην Ένωση σημαίνει ότι 50 δισεκατομμύρια χάνονται από τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών ετησίως. Είναι πολλά τα χρήματα αυτά και χρειάζονται ένα μεγάλο μηχανισμό ξεπλήματος. Αντίστοιχο με αυτό που είδαμε στα έγγραφα του Παναμά ή των φορολογικών παραδείσων. Πρόσφατα η Βουλή των Κοινοτήτων στη Βρετανία δημοσίευσε μια σχετική μελέτη για την απάτη ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο και κατέδειξε τα προβλήματα που έχει το σημερινό σύστημα και ζητάει να αναλυφθεί δράση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται ότι η απόλυση ήταν της τάξης του 1 με 1,5 δισεκατομμύρια ε, λίρες στερλίν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ποιε είναι τώρα οι πρωτοβουλίε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παίρνει πολύ στα σοβαρά υπόψη αυτό το θέμα. Ο πρόεδρο Γιούνκερ είπε ότι χρειάζεται μια πιο καλή εσωτερική αγορά που να λειτουργεί καλύτερα και αυτό είναι προτεραιότητα της θητείας του και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει οι εταιρείε να φορολογούνται ε, όσο τους αναλογούν. Τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που εφαρμόζουν τους κανόνες ΦΠΑ. Αυτό το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις φοροποφυγής. Ε, το είδαμε και στα διάφορα έγγραφα ε, το ΦΠΑ με διάφορους τρόπους ε, που αποκτούν κάποιοι θαλαμιγούς ή ιδιωτικά αεροσκάφη καταφέρουν να παρακάμψουν ε, το ΦΠΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει να γίνουν έρευνα. Όπως ε, ανέφερε και ο κύριος μάτε στο Συμβούλιο, ο Υπουργών Οικονομικών ΕΚΟΦΗΝ 22 Ιουνίου συμφώνησε μια, μια κοινή προσέγγιση μετά από πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε οι εθνικές εφορίε, να έχουν πιο αποτελεσματικά νέα έργα για να καταπολεμούν αυτό το θέμα της απάτης στο ΦΠΑ, να κάνουν κοινέ αναλύσεις κινδύνου και από κοινού να ανοιχνεύουν και να καταπολεμούν την οργανωμένη απάτη. Αυτή η νέα πρόταση επίσης επιτρέπει ε, να μοιράζονται δεδομένα και πληροφορίες με την Ευρωπόλ, την Όλαφ και τα τελωνία ε, για να ε, υπάρξει νομική βάση έτσι ώστε να προχωρούν στη δίωξη αυτών των υποθέσεων. Το θέμα είναι στο Κοινοβούλιο για γνωμοδότηση και Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων γνωμοδότησε ήδη τον Ιούνιο και περιμένουμε την τελική. Τρίτον, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι Ακόμα και αν έχουν ενισχυμένε δυνατότητε οι εφορίε για την καταπολέμηση του ΦΠΑ, το σημερινό σύστημα χρειάζεται ξεχρονισμό γιατί επιτρέπει απάτε. Γι' αυτό πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αλλάξει το σύστημα ΦΠΑ ε, σε ό,τι αφορά τους, ε, τις ενδομιλικές ε, συναλλαγές ή τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει αυτό, ότι Κάποιος που παρέχει ε, αγαθά και συλλέγει ΦΠΑ από ε, τον πελάτη του θα πρέπει να το καταβάλει. Έτσι θα μειωθεί ε, κατά 40 δισεκατομμύρια ετησίως η φορολογική απάτη με το ΦΠΑ. Αυτή είναι η δική μας πρόθεση, έτσι ώστε να ε, περάσουμε από το σημερινό μεταβατικό προσωρινό σύστημα σε αυτό που ονομάζουμε οριστικό. Οι νέοι κανόνες θα συνδυαστούν με εισαγωγή τουλάχιστον στην πρώτη φάση της έννοιας ε, του ε, πιστοποιημένου φορολογούμενου. Δηλαδή είναι ένας φορολογούμενος που τον αναγνωρίζει η εφορία ως φυσικό πρόσωπο. Και μόνο σε αυτή την περίπτωση ε, θα μπορεί ε, ένα εμπόρευμα να περνάει σύνορα χωρίς να έχει καταβληθεί ΦΠΑ. Το ενδοκινοτικό εμπόριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2017 ενέκρινε μια νομοθετική πρόταση η οποία μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει τις βασικές αρχές ε, του οριστικού συστήματος όπως είπα, είναι η αρχή της ε, χώρας ε, προορισμού ε, και η μοναπευθυντική θηρίδα για την δήλωση ΦΠΑ. Έτσι θα το σύστημα πιο απλό και θα αντέχει στις απάτες. Αυτή η πρώτη πρόταση είχε και συνέχεια. Ήρθε η πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 25 Μαΐου για μια οδηγία που περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες και τις τεχνικές εφαρμοστικές διατάξεις για την ε, πρακτική ε, εφαρμογή του οριστικού καθεστώτος ε, συστήματος. Ελπίζουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να δώσουν συνέχεια και γρήγορα, γιατί το θέμα είναι επίγον. Ολοκληρώνοντα, θέλω να σα πω ότι η καταπολέμηση απάτη είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα πρέπει να δούμε τη δυνατότητα των εφοριών να ε, επιβάλλουν αυτού του κανόνε και να συνεργάζονται για να ε, πατάσετε η απάτη στο ΦΠΑ. Αλλά και το ίδιο το σύστημα. Ήταν χρήσιμες οι διοικητικές ε, πρωτοβουλίες για να κλείσουν τα παραθυράκια και τα ελλείμματα, αλλά δεν αρκούν. Θα πρέπει να υπάρξει ένας εξυγχρονισμός έτσι ώστε να ευθυγραμμιστεί πλήρως το σύστημα ΦΠΑ στην εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και προσβλέπω στη συζήτηση που θα γίνει στη συνέχεια. Σα ευχαριστούμε για αυτή την άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα στην φορολογική αρχή τη Σουηδία, η κυρία Άλμα Ολαυστότηρ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε μέλη της Επιτροπής ε, τα 3. Ευχαριστώ που καλέσατε σε αυτήν την ακρόαση για να συζητήσουμε την διασυνοριακή απάτη του ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρχικά θα ήθελα στην παρουσίασή μου να παρουσιάσω τον ρόλο του δικτύου Eurofisk στην καταπολέμηση της απάτης ΦΠΑ και ιδίω την ε, απάτη, την κυκλική απάτη ενδοκινοτικά, την απάτη του αθανούς εμπόρου που ονομάζεται και MTIC Πρέπει να πω ότι η απάτη αυτή ειδικά του αφανούς εμπόρου έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες και έχει γίνει μείζον πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα συστήματα εξαπάτησης γίνονται ολένα και πιο περίπλοκα και εξαπλώνονται σε διαφορετικές αγορές. Είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς το ακριβέ ποσό απολειών από το ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά υπολογίζεται σε περίπου 50 δις ευρώ εξαιτία του ΦΠΑ ετησίω. Εκτίμηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι λοιπόν ζωτική σημασία η απάτη ΦΠΑ να προλαμβάνεται, να ανοιχνεύεται και να καταπολεμάται όσο το δυνατόν συντομότερα. Η απάτη του αφανού εμπόρου κυκλικής μορφή, μορφής ε, αφορά συνήθως ε, διαφορετικά συστήματα εξαπάτησης σε διαφορετικά κράτη-μέλη και μπλέκονται ε, πολλές φορολογικές αρχές από απαιτείται διεθνή συνεργασία. Το δίκτυο Eurofisk ιδρύθηκε βάσει του κανονισμού του Συμβουλίου 904 το 2010 για να ενισχυθεί η διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στην καταπολέμηση της οργανωμένης απάτης ΦΠΑ και ιδίω της κυκλικής απάτης του αφανούς εμπόρου. Η Eurofisk είναι ένα δίκτυο γρήγορη ανταλλαγή ε, στο στοχευμένο πληροφοριών μεταξύ των 100 μελών. Και τα 28 κράτη-μέλη συμμετέχουν στο δίκτυο, αλλά μπορούν να επιλέξουν σε ποιο τομέα του ενδιαφέρει να συμμετέχουν περισσότερο και πότε θέλουν να λήξει η συμμετοχή του. Όταν ε, συμμετέχει σε ένα τομέα εργασία, ένα κράτο μέλο υποχρεούται να συμμετέχει ενεργώ όπω έχει συμφωνηθεί από του υπόλοιπου συμμετέχοντε. Ε, αυτό έχει να κάνει με την φόρτωση ε, στοιχείων από και προς το δίκτυο Eurofisk και επίσης την ε, αντίδραση της πληροφορίες που λαμβάνει ο καθένας. Κάθε κάτω μέλος έχει ορίσει τουλάχιστον έναν υπάλληλο αξιωματικό σύνδεσμο, όπως θα λέγαμε, για τα θέματα τα φορολογικά που μπορεί να έχει εξειδίκευση στα θέματα του ΦΠΑ με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σε σχέση με διάφορες ε, περιοχές απάτης, ε, απειλές σε εθνικό επίπεδο, ε, τομείς κινδύνου και σχετικές πληροφορίες οι πληροφορίες στο δίκτυο ανταλλάσσονται μεταξύ των ε, υπευθύνων οπαλλήλων του Eurofisk και κάθε κράτος μέλος διορίζει έναν ε, συγκεκριμένο υπάλληλο για το δίκτυο Eurofisk και επίσης αυτός ψηφίζει εκπροσωπώντας το κράτος μέλος του στις διάφορες συνεδριάσεις του Eurofisk. Αυτή τη στιγμή το δίκτυο αποτελείται από την ομάδα Eurofisk και όσου εργάζονται σε διάφορους τομείς εργασία. Ο ρόλος της ομάδας, μεταξύ άλλων, είναι να αποφασίζει για τη δημιουργία και την πάυση λειτουργίας κάποιων ε, τομέων εργασία όπως λέγονται, και να αποτιμά τα αποτελέσματα του Eurofisk. Ο πρόεδρος εκλέγεται μεταξύ των υπαλλήλων υπευθύνων για ε, το Eurofisk που συμμετέχουν από τα διάφορα κράτη-μέλη. Αυτό εξαρτάται, μάλλον αριθμό των ε, τομέων εργασία εξαρτάται από τι ανάγκε μα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν έξι στο Eurofish και κάθε συντονιστή για κάθε τομέα εργασία συνεννοείται με του αρμόδιου υπαλλήλου. Το 2010 καταρτήσαμε τους πρώτους τέσσερι τομείς για να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένε περιπτώσεις απάτη του ΦΠΑ για το φορολογικό εισόδημα από το ΦΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρώτος τομέας εργασίας είναι ε, ο τομέας καταπολέμησης τη απάτη του αφανούς εμπόρου για όλα τα αγαθά και τι υπηρεσίε. Ο δεύτερος τομέα εργασία είναι νέα μέσα μεταφορών, ε, οχήματα, σκάφη και αεροσκάφη. Ε, ο τρίτο τομέα εργασία είναι οι καταχρήσει, οι παραβιάσει του, ε, της τελωνικής δικασίας 42.00 και εκπρόσωποι των φορολογικών αρχών και των τελωνιακών αρχών των κατομελών συμμετέχουν στο 2 και στο 3. Στον τομέα εργασία 4. Ε, Αυτό ε, λειτουργεί κάπω σαν παρατηρητήριο, λέγοντα μυστικέ ε, πληροφορίε για τι νέε τάσει και τι εξελίξει στα μοντέλα που ακολουθούν για την εξαπάτηση εγκληματίε και τις τεχνικές και προσεγγίσεις για την καταπολέμηση της απάτης ΦΠΑ. Έπειτα, ε, οι 5 και 6 μισό 5 και 6, δημιουργήθηκαν το 2016 και 2017 αντιστοίχως. Λόγω της παγκοσμιοποίησης και των ε, ε, τεχνολογικών εξελίξεων, ε, διαρκώς οι αρχές αντιμετωπίζουν προβλήματα συλλέγοντας δινοριακά τα έσοδά τους από το ΦΠΑ. Το 2016 δημιουργήθηκε η ομάδα για την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώση για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, που έχει μεγάλη σημασία για τη διεθνή οικονομία. Η εξέλιξη αυτών των νέων business model της παγκοσμιοποίησης, των νέων πλατφορμών εμπόριου, αλλά και πληρωμών δημιουργεί δυσκολίε στι φορολογικέ αρχέ προκειμένου να εντοπίσουν νέε περιοχέ κινδύνου και μοντέλα εξαπάτηση στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Υπάρχει σοβαρό κίνδυνο οφηγή του ΦΠΑ και εξαπάτηση στον τομέα αυτό. Ο τομέα εργασία 6 δημιουργήθηκε το 2017 για την υλοποίηση της ανάλυσης ε, δικτύου συναλλαγών με στόχο να ε, υποστηρίξει την λειτουργία του Eurofish και να γίνει πιο αποτελεσματικό το δίκτυο. Το TNA θα δημιουργεί αυτόματα πληροφορίε που πρέπει να ανταλλάσσονται και στο Eurofish και ώστε να βελτιωθεί η δυνατότητα των κρατών να αποστέλουν έγκαιρη προειδοποίηση και να αντιδρούν εγκαίρω με ποιότητα, αξιοπιστία, ασφάλεια ω προ τι πληροφορίε που ανταλλάσσουν. Το δίκτυο αυτό επιτρέπει να έχει κανείς μια σαφή εικόνα των δικτύων φορολογικής κυκλικής φορολογικής απάτης και μπορεί να επιταχύνει την ανείχνευσή τους. Θα αρχίσει να λειτουργεί πριν το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Το Eurofisk έχει αναμφίβολα συμβάλει στον περιορισμό των απολειών από το ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παρά τι προσπάθειε των 100 μελών να καταπολεμήσουν αυτή την απάτη και τη στενή διεθνή συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών, το πρόβλημα έχει ακόμα μεγάλη έκταση ε, και σοβαρέ διαστάσει λόγω της, του περίπλοκου χαρακτήρα και τη ταχύτητα με την οποία αναπτύσσονται οι τεχνικέ εξαπάτηση και οι νέε αγορέ. Οι μαζικές απώλειες μπορεί να πλέξουν και την αξιοπιστία της αγοράς, αλλά ακόμη και να συμβάλλουν στον αθέμητο ανταγωνισμό. Ας πούμε η αγορά ανταλλαγή δικαιωμάτων εκπομπών είχε πληγεί από την κυκλική απάτη το 2009-10 με απώλειες 5 δις από ΦΠΑ μόλις σε 18 μήνες. Και αυτό μετά επεκτάθηκε και στην αγορά ηλεκτρονικής ενέργειας και φυσικού, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Ε, άλλες αγορές όπως τα ηλεκτρονικά μέταλλα, ε, τηλεπικοινωνίες έχουν επίσης πληγεί και αυτό αφορά και αγαθά που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από εξωευρωπαϊκέ χώρες. Εξαιτία της διαδικασίας, διαδικασία 42.00 αλλά και των ε, συναλλαγών ε, εισαγωγών-εξαγωγών αυτό απαιτεί ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των ελληνικών αρχών, εξωευρωπαϊκών χωρών και όσων ε, δραστηριοποιούνται στην αγορά και τι επιχειρήσει. Παρά τις διάφορες προσπάθειες στα διάφορα κράτη-μέλη να καταπολεμήσουν την απάντηση του ΦΠΑ και τη διεθνή συνεργασία, υπάρχουν ακόμη δυσκολίες. Πολλά κράτη-μέλη έχουν προβλέψει συγκεκριμένε διαδικασίε αντιστροφή του βάρου τη ευθύνη τα τελευταία χρόνια και στα αγαθά και τι υπηρεσίε που συχνά έχουν να κάνουν με την εξαπάτηση του εθνού εμπόρου. Ε, ξέρουμε ότι κάπω περιορίζονται οι απόλυε από την απάτηση στο ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμω ε, η αντιστροφή του βάρους απόδειξης ε, δεν αρκεί. για την μετατόπιση της απάτης, γιατί μπορεί πολύ εύκολα κάποιος να περάσει την απάτη σε ένα άλλο κάτω μέλος ή σε νέες αγορές. Συνήθως οι φορολογικές αρχές που είναι υπεύθυνε για την αποτίμηση και τη συλλογή των εσόδων από το ΦΠΑ και παίζουν ε, καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη και την ανείχνευση της φορολογικής απάτης. Οι πληροφορίες των ε, φορολογικών αρχών όπως φτάνουν στο δίκτυο και είναι απόρριτες βάσει του άρθρου 55 του Συμβουλίου του συμβουλιου 904-2010. Δηλώνεται ότι οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται θα καλύπτονται από την υποχρέωση του επαγγελματικού απορρίπτου και η προστασία τους ε, καθορίζεται, επεκτείνεται και βαρύνει και το κράτο μέλος που τις λαμβάνει. Και αυτό αλλάζει ακόμη και για τις, μάλλον μπορεί να γίνει ακόμη και για τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται στα πλαίσια ποινική ε, έρευνα, ποινική δίωξη. Θα πρέπει βεβαίως οι διεκτικέ αρχέ ενό κράτου μέλους ε, να μπορέσουν να ε, ανταλλάξουν τι πληροφορίε ελεύθερα ανάλογα με του κανόνε των κρατών μελών σε περίπτωση που χρειάζεται συνεργασία. Ο ορισμό του οργανωμένου εγκλήματο ε, και των εγκληματικών ε, ομάδων είναι διαφορετικό. Βρίσκεται σε πολλά, μάλλον επίσημα ευρωπαϊκά έγγραφα. Η, απάτη του, η κυκλική απάτη του αφανού εμπόρου είναι σοβαρό δίκημα και διαπράτεται από εγκληματικέ ομάδε. Βάσει των στοιχείων τη Europol, 40-60 δι ευρώ είναι οι αιτήσιε απώλειε από το εισόδημα του ΦΠΑ λόγω τη δράση των ομάδων αυτών και 2% έχουν να κάνουν ακριβώ με το 80% των απατών αφανούς εμπόρου. Αυτό βεβαίω ε, καταλήγει και στη χρηματοδότηση τη νομοκρατία και έχει να κάνει και με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο. Έτσι λοιπόν, όλοι οι φορεί και το δίκτυο που είναι υπεύθυνο για την καταπολέμηση τη απάτη του αφανού εμπόρου πρέπει να συνδυάσουν τι δυνάμει του σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για να βρούμε περισσότερε ευκαιρίε να αναχαιτήσουμε αποτελεσματικά την κυκλική απάτη του εμπόρου και του ΒΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να περιορίσουμε τις φορολογικές ε, απώλειες, αλλά και να προσάγουμε στη δικαιοσύνη τη υπεύθυνη ομάδα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τώρα ο κύριο. Μάφη, ευχαριστώ πολύ. Έχω κάνει έρευνε για το θέμα αυτό. Ε, στα πλαίσια ενός προγράμματος του Ορίζοντα 2020 που λέγεται καταπολέμηση της ε, απάτης και ε, ενίσχυση των ρυθμιστικών αρχών. Και κοιτάζω τα θέματα αυτά από πιο μακροοικονομική αρχή και χαίρομαι που ε, δεν θα αναφέρω τα θέματα τα οποία θα αναφέρετε εσείς και επειδή κάποια θέματα καλύφθηκαν θα μιλήσω λίγο διαφορετικά. Γιατί δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα με ρωτήσατε και νομίζω πως είναι σημαντική ερώτηση. Ένας από τους λόγους είναι ότι δεν αλλάξαμε ακόμη την νομοθεσία για το ΦΠΑ και ακούσαμε ήδη ότι είναι σε φάση αλλαγή, Ούτω ώστε να είναι με βάση τη χώρα ε, προορισμού. Νομίζω ότι τα νούμερα που αναφέρατε είναι απόλυτα σωστά γιατί ένα μεγάλο τμήμα των 50 δισεκατομμυρίων που χάνουμε θα καλυφθεί έτσι. Αλλά άκουσα επίση ότι η απώλεια ΦΠΑ μπορεί να είναι μεταξύ 125 και 150 δι. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Και αν το βασίσουμε αυτό στο μέγεθος της παραοικονομίας θα μπορεί να ήταν 135 δις. Δηλαδή κάπου εκεί κινούνται όλες οι εκτιμήσεις. Άρα και αν λύσουμε αυτό το πρόβλημα θα παραμείνει σημαντικό ποσό απάτης. Και αν κοιτάξω τα στοιχεία του Ηνωμένου Βασιλείου που νομίζω ότι έχει τα καλύτερα στοιχεία για την απώλεια ΦΠΑ ενώ έχει πολύ μικρή ε, παραοικονομία με βάση την Ευρώπη 62% των απολειών έχουν να κάνουν με την ε, ε παραοικονομία. 10% είναι με απομακρυνές ε, ε, ε πωλήσει, 13% είναι λόγω κακού χρέους και μόνο 4% είναι εγκληματική δραστηριότητα. Και είναι τόσο χαμηλό που σκεφτόμαστε να μην το αναφέρουμε στο παρελθόν και μόνο 1% είναι αποφυγή του ΦΠΑ. Εγώ είμαι ορκωτός λογιστής και χαίρομαι που δεν είμαστε πολύ παρόντος σε αυτό το τομέα. Το μεγάλο θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν είναι η παραοικονομία. Και αυτό είναι κυρίως ε, θέμα εσωτερικό, όχι διεθνές. Γιατί δεν έχουμε λοιπόν καλύψει τις απώλειες ΦΠΑ, γιατί ακριβώς, όπως και για πολλά άλλα φορολογικά θέματα τα τελευταία 15 χρόνια, από τότε που έγινε κύριο θέμα η φορολογική δικαιοσύνη, κοιτάξαμε την διεθνή διάσταση του θέματος, αλλά να θυμηθούμε ότι η εσωτερική διάσταση του θέματος αυτού είναι πολύ σημαντική για κάθε χώρα και νομίζω ότι το έχουμε υποτιμήσει. Αν εξετάσουμε τη σχετική σημασία που αποδίδουν τα κράτη-μέλη σε αυτό το θέμα, είναι απογοτευτικό ότι μόνο 14 από τα 28 κράτη-μέλη έχουν οποιαδήποτε εκτίμηση των ε, απολειών φόρων και οι περισσότεροι κυρίως εστιάζουν σχεδόν αποκλειστικά στον ΦΠΑ. Και όπως υπόθηκε, και από το Ελεκτικό συνέδριο έχουν μια προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω. Εγώ νομίζω ότι αυτή η προσέγγιση είναι η σωστή για το ΦΠΑ. Εγώ θεωρώ ότι όλα, όλες οι απώλειες φόρων πρέπει να υπολογίζονται με αυτόν τον τρόπο. Δεν αποκλείω και την προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, αλλά πιο σημαντικό είναι το αντίστροφο. Έχουμε μια εκτίμηση της Κομισιόν για την απώλεια ΦΠΑ συνολικά, αλλά αν τα κράτη-μέλη δεν αντιμετωπίζουν και στο εσωτερικό τους το θέμα αυτό, στη δική του οικονομία, από όπου προκύπτουν αυτέ οι απώλειε, τότε δεν καταλαβαίνω πώ μπορεί να έχουν αποτελεσματική στρατηγική αντιμετώπιση του θέματο αυτού. Γι' αυτό προτείνω στην Επιτροπή μα ότι θα πρέπει να συστήσει νομοθεσία που να λέει ότι όχι μόνο οι απώλειε ΦΠΑ, γενικά οι απώλειε φόρων πρέπει να υπολογίζονται από κάθε κράτο μέλο. Το λέω σαφέστατα αυτό. Γιατί αν χάνει πόρου από το ΦΠΑ, είναι φόρο επί του κύκλου εργασιών, ιδιαίτερα για την χώρα οικονομία και θα ξέρετε ποια είναι, ποιες είναι οι αρχές της λογιστικής. Εγώ είμαι ιδιαίτερα εξοικειωμένος. Εάν δεν ε, καταγράψεις το φόρο εργασιών, τότε δεν θα καταγράψεις και τους φόρους εισοδήματος, τις ε, συνεισφορές και τον εταιρικό φόρο που πρέπει να υπολογίσεις. Άρα το κόστος, αν χάσεις το ΦΠΑ, είναι πολύ μεγαλύτερο από τις απώλειες ΦΠΑ. Άρα τα κράτη-μέλη πρέπει να αντιμετωπίσουν σοβαρά το θέμα αυτό. Και δυστυχώς δεν το κάνουν μέχρι στιγμής. Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα. Επιπλέον, και κάτι που ενισχύει αυτό που ήδη είπα, καμία εφορία δεν μπορεί να αξιοποιήσει τα στοιχεία αν δεν έχει και τους πόρους και το προσωπικό για να λύσει τα θέματα αυτά. Άρα, εάν δεν έχουν επαρκείς πόρους οι φορολογικές αρχές, δεν κάνουμε τίποτα. Σε πολλές χώρες οι κυβερνήσεις θεωρούν ότι οι εφορίες ε, κοστίζουν αντί να φέρνουν εισόδημα. Δεν καταλαβαίνω αυτή τη λογική ως λογιστής και ως επιχειρηματίας. Εάν κάτι μου φέρνει χρήμα, μ' αρέσει. Αλλά εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να μειωθεί η φορολογική μας αρχή από πλευρά πόρων. Αυτό είναι ακατανόητο. Για να λύσουμε τώρα το θέμα στο εσωτερικό κάθε χώρα. Πρέπει να κάνουμε μερικά σημαντικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ας δούμε το μοντέλο της Πορτογαλίας, το οποίο είναι ότι θα πρέπει κάθε πώληση που ηλεκτρονικά να αποστέλλεται στις φορολογικές αρχές. Λειτουργεί αυτό. Έχω κάποιες ε, ε, επιφυλάξεις για την επιγραμμική καταγραφή των φόρων, αλλά η καταγραφή του κύκλου εργασιών είναι ουσιώδης. Μ' αρέσει έτσι το κίνητρο που δίδεται. Ότι δηλαδή επίσης κάθε απόδειξη είναι ένας λαχνός για ένα εθνικό λαχείο. Βλέπω ότι υπάρχουν κάποιε επιφυλάξει. Δεν δουλεύει. Καλά, δεν ξέρω. Εντάξει, αν με πείσετε, αλλά εγώ νομίζω ότι η, η ιδέα αυτή είναι καλή. Αλλά το πιο σημαντικό θέμα που πρέπει να εξετάσουμε είναι το θέμα είναι ότι έχουμε στην εθνική οικονομία πολλές απώλειες από αυτούς τους αφανείς εμπόρους, αλλά και διεθνώς. Δεν χάνουμε μόνο ένα τμήμα του κύκλου εργασιών στην ουσία ε, δεν υπάρχουν, δεν καταγράφονται πουθενά αυτοί οι αφανεί συναλλασσόμενοι. Στο Ηνωμένο Βασίλειο τουλάχιστον 400.000 εταιρείε το χρόνο δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση για τον εταιρικό φόρο, όπως απαιτείται από τον νόμο. Και ποτέ δεν δίνουν και πληροφορίες φυσικά για τους πραγματικούς δικαιούχους τους. Οπότε υπάρχει ένα τεράστιο κενό στο φορολογικό μας σύστημα. Τουλάχιστον 10% των εταιριών ποτέ δεν δίνουν προφορίες για τι συναλλαγέ του. Και από αυτέ οι μισέ ποτέ δεν θα ε, δώσουν τέτοια στοιχεία καθ' όλη τη διάρκεια τη ζωή του. Μπορεί να υπάρξουν για ένα διάστημα, μπορεί να έχουν συναλλαγέ και μετά να εξαφανιστούν και κανεί δεν θα μάθει τίποτα. Επίση έχουμε 5 εκατομμύρια αυτοαπασχολούμενοι. Τα εισοδήματά του είναι πολύ κάτω από το ελάχιστο εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει συστημική υποδήλωση των εισοδημάτων τους. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μια συγκεκριμένη περίπτωση που θα είναι εμφανής και ε, πολύκροτη για να τους πείσει να δηλώνουν. Πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα εθνικό ανταλλαγής πληροφοριών. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει αυτόματη ε, ανταλλαγή πληροφοριών με τους φορολογικούς παραδείσους. Αυτό το λέω εδώ και πολύ καιρό. Όμως δεν κάνουμε κάτι για το εσωτερικό των δικό μας οικονομιών το εσωτερικό των οικονομιών μα. Για παράδειγμα, μια τράπεζα στα νησιά Κέιμαν πρέπει να ενημερώσει το Ηνωμένο Βασίλειο εάν κάποιο πελάτη τη διαμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο και να στείλει πληροφορίε και για τι επιχειρήσει του. Αλλά αν έχει μια επιχείρηση στο Λονδίνο ένα άτομο, δεν υποχρεούται. Αυτό είναι απόλυτα παράλογο. Πρέπει το σύστημα αυτό που ήδη υπάρχει και για το οποίο υπάρχει αναγκαία υποδομή να εφαρμοστεί και στο εσωτερικό τη κάθε χώρα και να το επεκτείνουμε σε όλους τους εσωτερικούς λογαριασμούς. Όταν υπάρχουν ύποπτες συμπεριφορές, που σημαίνει ότι γίνονται κάποιες συναλλαγές. Και πρέπει επίσης να επεκταθεί και σε όλες τις εμπορικές πλατφόρμες στο ίντερνετ και τις πλατφόρμες πληρωμών, όχι μόνο δηλαδή τις εταιρείες που συναλλάσσονται επιγραμμικά. Οπότε όλοι θα γνωρίζουν ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να τους πιάσουν. Και από μελέτες στις ΗΠΑ αποδεικνύεται ότι όταν κάποιοι θεωρούν ότι είναι πολύ μικρή πιθανότητα ότι θα αποκαλυφθούν οι συναλλαγές τους, τότε 50 έως 60% μόνο 50-60% θα δηλώσουν την πηγή του εισοδήματό του, ούτε καν το ύψο, μόνο την πηγή. Αν θέλουν ότι η πηγή θα δηλώσει αυτόμητα, αυτόματα τους, ότι του ε, ε, παρέχει εισόδημα, τότε το ποσοστό αυτό ανέβει στο 90%. Η ανταλλαγή πληροφοριών στο εσωτερικό των οικονομιών θα μα βοηθούσε. Δεν χρειαζόμαστε πολλή πληροφόρηση. Οι τράπεζε πρέπει να μα δίνουν στοιχεία για του πραγματικού δικαιούχου. <clears throat> και ε, οι επιχειρήσει ακόμη στον Ηνωμένο Βασίλειο δηλώνουν ότι την άνοιγε και κανεί δεν ελέγχει. Θα πρέπει οπωσδήποτε οι τράπεζε να ελέγχουν του πραγματικού δικαιούχου, να ενημερώνουν τι ε, φορολογικέ αρχέ, ούτω ώστε να έχουν επαρκή στοιχεία για να βρούμε αυτού του αφανεί εμπόρου. Μόνο έτσι θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Και παράλληλα θα στηρίξουμε τους ε, εντύμους επιχειρηματίες των οποίων η ανταγωνιστικότητα μειώνεται όπως θα έπρεπε να είναι ο στόχος του εγχειρήματό μας. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μέρφη και όλους τους ομιλητές μας για τις εισαγωγικέ αυτές παρουσιάσεις. Αρχίζει η συζήτηση, όπως πάντα, ερωτήσεις. Ένα πεντάλεπτο κάθε ερώτηση, ένα λεπτό ερώτηση και το υπόλοιπο για τις απαντήσεις. Αν έχουμε χρόνο, μπορούμε να κάνουμε και δεύτερη ερώτηση, ευκρινιστική, συμπληρωματική. Ο κύριος Μάγερ, συνεισηγητής από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ και τους αγαπητούς ε, προσκεκλημένους που ήρθαν για να συζητήσουν μαζί μας αυτό το σημαντικό φορολογικό θέμα. Όπως ακούσαμε το πρωί, είναι και αντικείμενο εγκληματικών δραστηριοτήτων και άλλων ε, παράνομων ενεργειών. Είχα την αίσθηση και επιβεβαιώνεται από τη συζήτηση ότι το διασυνοριακό εμπόριο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και έχω και μια ερώτηση προς την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. θα είναι αποτελεσματική αυτή η αλλαγή του συστήματος ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειωθεί η απάτη. Κύριε Κόμες, εκπλήσεστε που υπάρχει τέτοια αντίσταση από τα κράτη-μέλη. Υπάρχει και πολύ μεγάλη έλλειψη εμπιστοσύνης ε, μεταξύ των κρατών και των φορολογικών αρχών. Πώς θα προχωρήσουμε. Ποιος να απαντήσει πρώτος στο ελεκτικό συνέδριο ή εσείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι, ο κύριος Μάτες. Για, αναφερθήκατε στο ευρωπαϊκό εμπόριο. Δεν είμαι βέβαιος ότι με την ηλεκτρονική δήλωση που ισχύει τώρα δεν είμαι βέβαιος ότι δεν, μπορεί να, δεν μπορούν να επιτευχθούν τα ίδια αποτελέσματα που επιθυμούμε. Αν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι αναφέρονται στο VIS όλες οι συναλλαγές, ιδιαίτερα οι εισαγωγές, είναι σαν να θες να δημιουργήσεις ένα σύστημα, πώς να το πω, Ε, όπου ψάχνεις τον τελικό δικαιούχο. Αυτό είναι εύκολο να βρεθεί από τη χώρα προορισμού και είναι εύκολο να συλλεγούν τα στοιχεία. Ξέρεις ποιος είναι ο τελικός αποδέκτης του προϊόντος. Ας πούμε, η εφορία σε μια χώρα μέλος Α ε, συλλέγει φόρους που μετά θα πρέπει να μεταβιβάσει στη χώρα Β, που είναι χώρα προορισμού αυτό δεν πρόκειται να το δεχθούν εύκολα. Και δεν είμαι βέβαιος ότι θα το δεχτούν οι χώρες που δικαιούνται να συλλέξουν αυτά τα έσοδα ή να τα εισπράξουν. Δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν θα υποτιμούσα τις ε, πολιτικές δυσκολίες. Υπάρχουν και πιο απλές λύσεις. Υπάρχουν ηλεκτρονικά στοιχεία από το σύστημα VIS και από τα τελωνία. Και υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί και με αποτελεσματικότητα. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα υιοθετηθεί έτσι εύκολα ένα σύστημα όπου κάποια φορολογικά έσοδα, ας πούμε, που δικαιούται η Γαλλία θα τα συλλέγει μια άλλη χώρα και θα τα μεταβιβάζει. Δεν είναι τόσο εύκολο. Τι γίνεται με το σημερινό σύστημα. Μπορεί να ενισχυθεί και δίδαση προς το σκέλος της επιβολής και της δίωξης ε, προσφέρεται για να ε, καταπολεμηθεί η απάτη στο ΦΠΑ. Αυτό ήταν το δικό μου σχόλιο. Ευχαριστώ. <laughs> Σίγουρα αυτό θα πυροδοτήσει και κάποιες άλλες σκέψεις. Η κυρία Ολαυστοτήρ. Α, όχι. Δεν θέλετε εσείς. Ο κύριος Μέρφυ. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Πρέπει να αλλάξει το σύστημα ΦΠΑ. Ε, απλή απάντηση. Για τη δεύτερη ερώτηση και την πολιτική βούληση, όπως αναφέρετε κι εσεί. Πριν από λίγα χρόνια, ε, διάβασα ένα βιβλίο που λεγόταν The Joy of Tax, η χαρά του φόρου, που δεν ε, συμφωνούσαν όλοι. Αλλά το θέμα ήταν η πολιτική βούληση. πώς μπορεί ένας πολιτικός να διαμορφώσει, να διαμορφώσει την οικονομία για την οποία είναι αρμόδιος. Αλλά αυτοί το χρησιμοποιούν για τους πολιτικούς σκοπούς. Δυστυχώς ακόμα πολλοί πολιτικοί θεωρούν τη φορολογία ε, ως εμπόδιο, κατάσχεση ή οτιδήποτε. Πρόκειται για ένα ε, στοιχείο περιουσιακό του κράτους ε, που συλλέγεται και αποδίδεται. Ε, δεν πρόκειται οι πολιτικοί, πιστεύω, να ανταποκριθούν ε, έτσι, με ενθουσιασμό να πούν ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Μάλλον καταστολή της αγοράς, το θεωρώ. Ευχαριστούμε, κυρία Ολαυστότηρ. Θέλετε? Όχι, Επιτροπή. Ναι, να απαντήσω στην ερώτηση που απευθυνόταν συγκεκριμένα στην Επιτροπή για το συγκεκριμένο καθεστώς και τις ε, ιδέες που παρουσίασε το περασμένο Οκτώβριο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πρώτες αντιδράσεις στο Συμβούλιο ήταν να συμφωνήσουν μόνον επί της αρχής, χωρίς να ε, γνωρίζουν τις λεπτομέρειες βέβαια. Αυτό ήταν δύσκολο Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε γρήγορα για να δώσει και τις λεπτομέρειες. Τις λεπτομέρειες προκειμένου να μπορεί να εφαρμοστεί όλο αυτό με τα stones, στα σημεία ορόσημα που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Για την έλλειψη εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών όπως την έθεσε ο κύριος Μάτος και για, τον, για την εννέα θηρίδα, εδώ μπορούμε να πούμε ότι το, η μήνυ εννέα θηρίδα ήδη λειτουργεί για κάποιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και βάσει των πληροφοριών που λαμβάνουμε από τα κάτι μέλη, χαίρονται πολύ. Τους αρέσει το σύστημα. Διότι τώρα επιτέλους παίρνουν χρήμα που πριν το χάνανε από αυτές τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Τον Δεκέμβριο το Συμβούλιο συμφώνησε επίσης το πακέτο ε, ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η ενιαία θηρίδα θα καλύπτει πλέον ε, και άλλα πτυχές του ηλεκτρονικού εμπορίου. Υπό αυτήν την έννοια ξέρουμε ότι είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών μελών και ένα από τα μέτρα που θα μας το επιτρέψει αυτό είναι η κοινή έλεγχη. Τα κάτι μέλη συμφώνησαν στο ΕΚΟΦΗΝ την περασμένη Παρασκευή να διοργανώνουν κοινού ελέγχου. για να μπορούν να γίνουν ε, κοινοί λογιστικοί έλεγχοι. Αυτό είναι ένα πρόσθετο βήμα και πέραν αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρχίσει τις συναντήσεις με τους διευθυντές των φορολογικών αρχών των κρατών μελών. Μια πρώτη συνάντηση έγινε πριν από λίγες μέρες και σε λίγες, μέρες, εβδομάδες θα έχουμε συνάντηση πάλι στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα. Όλοι οι διευθυντές των εθνικών φορολογικών αρχών συνεργάζονται και βρίσκονται για να συζητήσουν ε, τα ζητήματα που τους απασχολούν. Είναι αυτό ένα ξεκίνημα για να αρχίσει να υπάρχει εμπιστοσύνη κάτι που είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε τελικά να δημιουργήσουμε έναν ενίο ευρωπαϊκό χώρο του ΦΠΑ. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Κόφοδ, ε, εισηγητής για τους ε, σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους ε, συμμετέχοντες για τις παρουσιάσεις τους. Έχω μια ερώτηση για όλους με αφορμή την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τον ΦΠΑ. το πιστο, ο πιστοποιημένος φορολογούμενος που έχει ε, οργανώσει η Επιτροπή και ισχύει και για εταιρείε και για την εξεπάτηση του αφανούς εμπόρου. Πώς αξιολογούν τα μέλη του πάνελ το μοντέλο αυτό είναι αποτελεσματικό για να καταπολεμήσουμε την απάτη του ΦΠΑ και αν όχι μπορούμε να το βελτιώσουμε. Και επειδή τα κράτη-μέλη εδώ είναι πολύ επιφυλακτικά Εάν το μοντέλο αυτό δεν εφαρμοστεί όπως προβλέπετε, τι άλλες εναλλακτικέ υπάρχουν για την καταπολέμηση της απάτης ΦΠΑ. Και εσείς κύριε Μέρφη, για την καταπολέμηση της απάτης ΦΠΑ είπατε ότι ίσως ηλεκτρονική εγγραφή των εμπορικών συναλλαγών που να γνωστοποιούνται αμέσως της φορολογικής αρχής να ήταν μια πρώτη λύση. Αυτό εμένα μου δημιουργεί κάποιες αμφιβούλειες. Ίσως για άλλες φορολογικές απάτες αυτό το σύστημα ήταν αποτελεσματικό γιατί από το μέρισμα των φορολογικών απατών στην Ευρώπη βλέπουμε, λόγω χάρη μεταξύ δανέζικων και γερμανικών αρχών, να έχουν εντοπιστεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε απώλειες. Ε, αυτό θα μας ενδιαφέρε. Ευχαριστώ. Για την πρώτη ερώτηση. Καλά, ξεκινήσουμε απευθείας από τον κύριο Μέρφη με τη δεύτερη ερώτηση. Εάν θέλετε να απαντήσω στη δεύτερη αλλά και στην πρώτη εντάχει. Μου αρέσει η ιδέα του μοντέλου CTP. Ανησυχώ βεβαίω ότι θα πρέπει κανείς να αποδείξει σε ποιο καθεστώς εγγράφεται και αυτό είναι ένας πρώτος φραγμός για την είσοδο στην αγορά. Ίσως οι κυβερνήσεις πρέπει να αναζητήσουν τρόπους ώστε να δώσουν στήριξη στις μικρές επιχειρήσεις που θέλουν να, να μεγαλώσουν, να αυξήσουν τη δραστηριότητά του για να μην τους γύρει φραγμούς. Από την πλευρά του ψηφιακού μερίσματος. Πώς γράφεται κανείς δεν είναι το πρόβλημα, το blockchain, οτιδήποτε άλλο. Αυτό που μετράει είναι ακριβώς, δεν είναι καν ούτε οι συγκεκριμένε λεπτομέρειες. Είναι να γνωρίζει κανείς ότι υπάρχει ροή πληροφορίας. Έχει να κάνει όλο αυτό με το πώς συμπεριφερόμαστε από οικονομικής σκοπιάς, όχι με τις λεπτομέρειες. Δηλαδή στις τράπεζες ε, ή στις επιχειρήσεις θα έπρεπε να δούμε πού γίνονται οι συναλλαγές και πού γίνονται οι πωλήσει των συγκεκριμένων επιχειρήσεων με καταγραφή των σημείων πωλήσεων. Αυτά ε, μπορούμε να τα γνωρίζουμε. Σίγουρα θα υπάρχει περιθώριο σφάλματο, διότι άλλοι προτιμούν τα μετρητά, άλλε συναλλαγέ μέσω τραπεζικών λογαριασμών, ε, που μπορεί να μην έχουν σχέση με πωλήσει, να είναι ροέ κεφαλαίου ή μυρισμάτων που είναι άλλη μορφή έσοδα ε, και εκεί να χρειάζονται κάποιε επεξηγήσει. Αλλά το γεγονό ότι κάποιο γνωρίζει ότι υπάρχει υποχρέωση, υπάρχει νομικό περιορισμό, αυτό αντιστρέφει την ε, υποχρέωση λογοδοσία και του ε, αναθέτει τον ρόλο, την ευθύνη ε, της απόδειξη. Αυτό υποχρεώνει του τους λογιστές και όλους όσοι κινούνται γύρω από μια επιχείρηση να προσαρμοστούν όχι στο, τι ίσχυε πριν από 20 χρόνια αλλά να τους πούν ε, κάνε αυτό που πρέπει γιατί θα έρθει κάποιο και θα σε, θα περιλάβει. Ε, και ήταν πιο ευχάριστη η προσέγγιση που επέτρεπε ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Ε, αλλά Προ στιγμήν η λογιστική έλεγχη ΦΠΑ στις χώρες, ε, στις διάφορες χώρες είναι πολύ περιορισμένη και αυτό είναι μια δυναμία μα για τα ψηφιακά λοιπόν πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα, συγκεκριμένε υποχρεώσει. αν γνωρίζουμε ποιο είναι αυτό που εμπορεύεται μπορούμε να εντοπίσουμε που είναι και ο κίνδυνο, διότι η διαφορά μεταξύ τη ε, εξωτραπεζικής δραστηριότητας και της τραπεζικής είναι το πρόβλημα το πώς ε, μπορεί ο καθένα να έρχεται κοντά προ του δείκτε και να φαίνεται ότι συγκλίνει είναι ένα πρόβλημα. Εγώ ήμουν υπέρ τη άποψη να υπάρχει υποβολή εκθέσεων ανά χώρα. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ε, πολυεθνικές να γνωρίζουν ότι επειδή είναι, ε, υπάρχει περίπτωση να ελεγχθούν, να προσέχουν διαφορετικά. Αυτό θα ίσχυε και για όλες τις επιχειρήσεις. Ευχαριστούμε. Η ε, κυρία Φάβραγκας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, για το CTP, για το καθεστώς αυτό, το θέμα είναι ότι θα υπάρχει ευθύνη του προμηθευτή. Εκτός, όπως είπα, εάν ο πελάτης είναι CTP, δηλαδή είναι κάποιος ε, πιστοποιημένα ε, αξιόπιστος ε, πληρώνει αξιόπιστα το φόρο του και είναι σαφές ότι θα πληρώσει τον, ε, και το ΦΠΑ στη χώρα προορισμού. Έχουμε τώρα αυτή τη νέα έννοια. για να διευκολύνουμε την μετάβαση προς την αρχή της χώρας προορισμού. Και μια άλλη ερώτηση για το CTP. Θα βοηθήσει την καταπολέμηση της ναι, γιατί είναι ένας αξιόπιστος ε, φορολογούμενος. Θα πληρώσει τον ΦΠΑ που του αναλογεί. Υπάρχει κίνδυνος αν δεν μπει στην οδηγία, στην πρόταση. Όπως είπα, είναι μετάβαση προς το πλήρες τελικό καθεστώς. Τώρα θα το εξετάσουν τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο για να δουν εάν χρειαζόμαστε αυτό το ενδιάμεσο στάδιο, θα λειτουργούμε με CTP. Ή αν θα παραμείνει αυτό το χαρακτηριστικό και στο τελικό καθεστώς. Ή αν μπορούμε να περάσουμε στην ε, αρχή του προορισμού και το, την ευθύνη του προμηθευτή. Χρειαζόμαστε και στοιχεία. Θα δούμε αν θα μπορέσουμε να ε, συμπεριλάβουμε το πιστοποιημένο υποκείμενο στο φόρο, αλλά φυσικά το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη θα δούνε ποια είναι η πιο κατάλληλη προσέγγιση. Ο κύριος Τόμ Φάντεν Κάντελαρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλημέρα σας. Αγαπητοί παρόντες σας πω και ζητώ συγγνώμη που δεν ε, μπόρεσα να είμαι παρόν στις παρουσιάσεις σας. Έρχομαι από άλλη επιτροπή. Διάβασα όμως τις απαντήσεις σας. Και ε, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι για το κόστος ε, συμμόρφωσης στο ΦΥΠΙΑ. Στο Βέλγιο, κατά μέσο όρο, πληρώνει μια εταιρεία 27.500 ευρώ για να προσαρμοστεί και να συμμορφωθεί στο περίπλοκο σύστημα ΦΠΑ που έχουμε. Πάνω από 50% του κόστους είναι η ειδική συμμόρφωση προς το ΦΠΑ. Ε, τήρηση βιβλίων ΦΠΑ, προετοιμασία και δήλωση ΦΠΑ, ε, πληροφορίες για τα διάφορα συστήματα ΦΠΑ στα κράτη-μέλη. Και είναι υψηλότερο το κόστος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εγώ εργάζομαι σε αυτό το θέμα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Είναι σημαντικά υψηλότερο το κόστος ε, για τις μικρομεσαίες σε σύγκριση ε, με τις πολυεθνικές. Αν είναι μια εταιρεία μέχρι 50 ε, εργαζομένους, ε, πληρώνει το 0,75% για αυτό, ενώ για τις μικρομεσαίες που έχουν μέχρι 20 υπαλλήλους είναι 7,4%. Λοιπόν, είναι τεράστιο το κόστος για τη συμμόρφωση στο ΦΠΑ. Βεβαίως υπάρχει ένας, ε, και ένα αντάλλαγμα ε, σε αυτά. Ε, σας είπα ότι είναι πάρα πολύ περίπλοκο και συγκεκριμένο το σύστημα και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μάτες και τον κύριο Μέρφη. Χρειάζονται περισσότερη έλεγχη ή να προσπαθήσουμε να απλουστεύσουμε το σύστημα το ΦΠΑ και προς την κυρία Φάμπρεγας. Πώς θα καταπολεμήσετε τη μη συμμόρφωση προς το ΦΠΑ ε, για τις προπληρωμές, για την ε, δήλωση σε πραγματικό ε, φόρο και πάει λέγοντας. Αλλά είναι πάρα πολύ περίπλοκες όσο και δαρπανήρες όλες αυτές οι δικασίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς βλέπει στο μέλλον τη λύση ε, και έχετε έτσι μια γενικότερη θεώρηση ή απλώς κάποια στοιχεία που τα προσθέτετε και τα συνενώνετε σε μια πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ο κύριος Μάτερ. Η εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για το ΦΠΑ θα βοηθήσει. Αν κάθε επιχείρηση πρέπει να εφαρμόσει την αρχή της χώρας προορισμού, επειδή είναι τόσο διαφορετική η νομοθεσία από πολλέ σημαντικές πλευρές για το ΦΠΑ των κρατών μελών θα είχε τεράστιο κόστος συμμόρφωσης. Κάποια εναρμόνιση θα βοηθήσει λοιπόν πολύ και θα συμβάλλει από πολλές απόψεις στη μείωση των ευκαιριών για απάτες υπήρχε η πρόταση να ενιοποιηθούν στοιχεία για τον τρόπο πληρωμής του ΦΠΑ. Να εναρμονιστεί τουλάχιστον η δήλωση για τον ΦΠΑ. Και απέτυχε. Άρα ε, καταλαβαίνετε πιο φιλόδοξα εγχειρήματα δύσκολα θα επιτύχουν. Αλλά φυσικά η εναρμόνιση του ΦΠΑ θα ήταν ένα τεράστιο βήμα πρόοδου. Αυτή, αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση. Ο κύριος Μάφη. Τώρα ούτε μπορώ να θυμηθώ πόσες δηλώσεις ΦΠΑ έχω κάνει για μένα ή για τους πελάτες μου. Πάρα πολλές. Δεν νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό αυτό το 27.000. Είναι ρεαλιστικό, είναι υπερβολικό. Κάθε χαρτί που γράφει ΦΠΑ, ούτως ή άλλως, για λογιστικού λόγους πρέπει να το επεξεργαστείς. Άρα το συμπληρωματικό κόστος για ε, αυτήν την επιπλέον συμμόρφωση είναι τόσο ακριβή. Βέβαια μπορεί να γίνουν λάθη. Ένα απλούστρο καθεστώ για μικρομεσαίε θα βοηθούσε. Αλλά δυστυχώ η πείρα από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ότι γίνεται κατάχρησή τους και χρησιμοποιούνται για απάτες. Άρα τελικά τα έχουμε καταργήσει. Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ενιαίο συντελεστή για τις μικρές επιχειρήσεις. Αλλά και αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί για απάτες. Ναι, ούτως ή άλλως για το ΦΠΑ είναι πολύ άδικο το ουσιώδες κόστος. Είναι ε, οι αυτόματες κυρώσεις ε, σε κάποιες χώρες αν κάνεις λάθος ή αν καθυστερείς τις δηλώσεις. Κάποιες μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν να προλάβουν ορισμένα πράγματα. Δεν υπάρχει καμία ανοχή αν αργήσει στην υποβολή. Και όλα τα λάθη, είτε καλόπιστα είτε όχι, τιμωρούνται αυστηρά. Αυτά είναι άδικα. Είναι κατά των αρχών της φυσικής δικαιοσύνης. Πρέπει οπωσδήποτε να διαχωριστεί από το θέμα της απάτης γιατί είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι, είναι βάρος και προκαλεί και φόβους στις μικρές επιχειρήσεις. Γιατί πραγματικά υφίστανται κυρώσεις. Το τονίζω λοιπόν αυτό. Να πλουστεύσουμε το σύστημα βεβαίως. Αλλά δεν ενθαρρύνω άλλες χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Όσοι είμαστε στην Ένωση όπου έχουμε πολύ υψηλό κατόφλι για την εγγραφή στο ΦΠΑ, γιατί αυτό δημιούργησε άλλα προβλήματα. Πολλές επιχειρήσεις δηλώνουν ε, κύκλο εργασιών ακριβώς κάτω από το κατόφλιο. Οι περισσότερε υποθέτω εντύμω, γιατί το κόστος υπέρβαση αυτού του κατοφλίου ε, τελικά είναι αντικίνητρο για να μεγαλώσει την επιχείρησή σου. Πρέπει να απλωστεύσουμε τι διαδικασίε για τι μικρέ επιχειρήσει. Αυτό είναι ο σωστό ε, Δρόμο για την επίλυση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το κόστος για τις μικρομεσαίες. Είναι υποσυζήτηση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μια πρόταση για να πλουστευτούν οι κανόνες για το ΦΠΑ για τις μικρομεσαίες. Και επιπλέον να τις βοηθήσουμε να λειτουργούν καλύτερα εντός της ε, ενιαίας αγοράς. Ο στόχος των προτάσεών μας είναι να απλουστευτούν οι κανόνες. Τώρα το κόστος ε, σε εθνικό επίπεδο, σε διάφορα κράτη-μέλη. Διαφέρουν τα συστήματα. Και αυτό μπορεί να επιφέρει πρόσθετο κόστος ή όχι. Όπως είπε και ο κύριος Μέρφυ, χρειάζονται βοήθεια κάποιες ε, επιχειρήσεις, όπως έχουν λάβει και για άλλα θέματα. Αυτό που έχουμε δύο στάσεις τάση στα κράτη-μέλη, όπως στην Ιταλία, την Ισπανία και νομίζω και στην Πορτογαλία και στην Ολλανδία και σε άλλα κράτη-μέλη, είναι ότι υπάρχει η τάση των εφοριών να ε, παρέχουν υπηρεσίες στους φορολογούμενους είτε μέσω πληροφορικής είτε μέσω ε, αυτομάτων συστημάτων ε, απαντήσεων σε ερωτήσεις, όλο και περισσότερο οι φορολογικές αρχές καταλαβαίνουν ότι πρέπει να συνομιλούν με τους φορολογούμενους. Όχι μόνο για να εισπράξουν τους φόρους, που φυσικά είναι ο στόχος ε, λειτουργίας των εφοριών, αλλά για να τους βοηθήσουν και να τους βοηθήσουν να συμμορφούνται με τους κανόνες. Αυτό διαπιστώνουμε ότι είναι τάση των εθνικών φορολογικών αρχών. Και οι προτάσεις μας ε, αφορούν το ΦΠΑ, αλλά σε εθνικό επίπεδο ο ΦΠΑ είναι μόνο ένας από τους φόρους που πρέπει να πληρώσουν οι εταιρείε. Οπότε εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν ασχολούμεθα με τον ΦΠΑ δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με το συνολικότερο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις φορολογικές υποχρεώσεις. Υπήρξε μια πρόταση να γίνει κάποια εναρμόνιση, όπως είπε και ο κύριος Μάτεν, αλλά δεν το δέχτηκαν τα κράτη-μέλη, αλλά έχουν περάσει χρόνια από τότε. Ίσως στο μέλλον να επιτύχουμε περισσότερη εναρμόνιση της συλλογής κάποιων φόρων. Αυτό θα βοηθήσει και τις εφορίες. Μέσω της βοήθειας που δίνουν για να ε, βοηθήσουν στους φορολογουμένους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ωραία. Σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο κύριος Κούν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω την ερώτησή μου στα γερμανικά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές και τις ομιλήτρες που ήρθα να απαντήσω στις ερωτήσεις μας. πρώτη ερώτηση απευθύνεται σε όλους και είναι μια ερώτηση επί της αρχής. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία των εθνικών φορολογικών αρχών με την Όλαφ. Γιατί σε κάθε, κάθε συζήτηση που είχαμε την Όλαφ εκφράζουν ε, τη λύπη τους ότι επικρατούν εθνικοί εγωισμοί Α πούμε η γερμανική εφορία έχει καλύτερε πληροφορίε και τι κρατάει για τον εαυτό τη. Και η Όλαφ, εντάξει, είναι καλή και την αγαπάμε, αλλά όχι και ως εταίρο για καταπολέμηση της απάτης. Και σας ρωτώ κύριε Όλαφ δάτια. Ε, η Όλαφ νομίζω δεν είναι τμήμα του δικτύου Eurofisk. Θα μπορούσατε να μας απαντήσετε πώς μπορεί να συμμετέχει. Και μετά, ερώτηση ιδιαίτερα προς τον κύριο Μέρφυ. Καταρχάς σας ευχαριστώ για την παρατήρηση ότι η εφορία δεν θα πρέπει να είναι ένας χώρος που θα πρέπει να γίνονται περικοπές και οικονομίες, αλλά μια υπηρεσία για να, ε, που να συλλέγει φόρους. Εγώ είμαι φοροτεχνικός και, και, και ξέρω περί τίνος ομιλείται. Ε, και μου είπαν ε, κάποιοι επισκέπτε ότι ε, στο παρελθόν στη Γερμανία η διαδικασία αντιστροφή της απόδειξη. Ε, ήταν καλό. Πώς μπορεί να διευρυνθεί για να καταπολεμήσουμε τη φορολογική απάτη στο φόρο κύκλου εργασιών και στο ΦΠΑ. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Στοτήρ, ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Όπως είπα και στην παρουσίασή μου, κάθε είδους συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και ε, ευρωπαϊκών ε, υπηρεσιών θα βελτίωνε τη δυνατότητα πάταξης της φορολογικής απάτης στο ΦΠΑ. Προς το παρόν, το Eurofisk είναι ένα δίκτυο μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών μελών κυρίω για να γίνεται μια ταχεία και ομαλή ανταλλαγή πληροφοριών. Εναπόκειται απολύτω στα κράτη-μέλη, όταν λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίε, ε, να διαθέτουν πόρους έτσι ώστε ε, να διεκπαιρώνουν αυτό το έργο και να μοιράζονται αυτές τις πληροφορίες με άλλα κράτη-μέλη. Ρωτήσατε αν μπορούν υπηρεσίε όπω η Olaf, η Europol να είναι τμήμα του δικτύου. Το θέμα δεν είναι τμήμα ενό δικτύου, γιατί ακόμα και αν είχε τη δυνατότητα το δίκτυο αυτό στο μέλλον να ανταλλάσσει πληροφορίες, ε, αυτό μπορεί να γίνει, αλλά χωρίς να είσαι και τμήμα του δικτύου. Σε ό,τι αφορά την αντιστροφή του βάρους της απόδειξης, Ε, όσα κράτη το έχουν εφαρμόσει αυτό, δεν είδα να σταματάει η απάτη. Ας πούμε στα κινητά τηλέφωνα 13 κράτη-μέλη ε, επέβαλαν το φόρο στον αποδεκτή και νόμιζαν ότι θα είχε τελειώσει η, η απάτη. Απλώς μετεγκαταστάθηκαν οι εταιρείες που κάνουν αυτές τις απάτες σε άλλα κράτη-μέλη. Γιατί φεύγουν εταιρείε και χάνουν και φορολογικά έσοδα από το ΦΠΑ οι χώρες που δεν εφαρμόζουν αυτό το είδος φόρου. Και οι συμμετέχουσες σε αυτές τις εταιρείες φεύγουν, πηγαίνουν αλλού. Δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, αν θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτός ο φόρος τον αποδέξει όλα τα κράτη-μέλη, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ευχαριστώ. Ο κ. Μέρφυ. Την πρώτη ερώτηση δεν μπορώ να τη σχολιάσω, δεν νομίζω ότι είναι στη δική μου αρμοδιότητα για το φόρο στον αποδέκτη. Ε, όταν εισήχθη ήμουν πολύ νέος τότε ε, για πρώτη φορά και αυτό έγινε για την καταπολέμηση της απάτης αλλά χρειάστηκε να εξηγηθεί πολύ αυτό στον κόσμο τι είναι αυτό και για ποιο λόγο το κάνουν. Και αυτό παραμένει. Γι' αυτό γίνονται όλες αυτές οι καταχρήσεις. Όλες οι καταχρήσεις στα λογιστικά προέρχονται από κάποιο είδος φραγμό, εμπόδιο όταν αλλάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς ενός προϊόντος ή ενός περιουσιακού στοιχείου. Ε, και πρέπει να βάλεις ένα σύνορο ή ένα όριο έτσι ώστε να καταγράφονται σωστά και από τις δύο πλευρές των σύνορων οι συναλλαγές. Και αυτό αφορά μια τεράστιο φάσμα, όχι μόνο το ΦΠΑ, ε, και όλη τη φορολογική απάτη και τους φορολογικούς παραδείσους και όλα τα συμπαραμαρτούντα. Για να κατανοούμε τι συμβαίνει κατέρωθα σε μια συναλλαγή. Το πρόβλημα είναι ότι ε, κάθε συναλλασσόμενος αν έχει διαφορετική μέθοδο εκεί χωράει και κατάχρηση και αυθαιρεσία. Και χρειάζεται κάποιο είδος διατησία Τώρα αν επεφέμεθα στην, στην τιμιότητα, υπάρχει πρόβλημα με το ε, θέμα της επιβολής φόρου στον αποδέκτη, αλλά ε, αν, ε, αν συλλέγεται σωστά ο φόρος προς τη θέμενης αξία, τότε ε, λύνεται αυτό το πρόβλημα, καταπίπτει και είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσετε. Μα αυτό στην αρχή το είχαν σκεφτεί ως λύση, όχι ως πρόβλημα. Ε, είναι μια προσωρινή λύση που δεν έλυσε το πρόβλημα αυτό, λέω. Ε, συμπληρωματική ερώτηση ο κύριος Κον. Ναι. Προς τον κύριο Μέρφυ επίσης, σωστά σας κατάλαβα ότι στο ε, Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχει εξωτερικός λογιστικός έλεγχος ε, των φορολογικών αρχών. Όχι. Όταν είσαι μεγάλη εταιρεία, μπορεί να έχεις κάποιον εφοριακό που να είναι στα γραφεία σου συνέχεια. Εμείς Για το ΦΠΑ δεν έχουμε στόχο αυτούς. Δηλαδή ε, η φοροαποφυγή, ε, οι μεγάλες εταιρείε δεν ε, έχουν φορολογική απάτη, έχουν φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Έγιναν μεγάλες περικοπές τελευταία δεκαετία στη Βρετανική εφορία και ο αριθμός των επισκέψεων έχει μειωθεί σε εμπόρους που είχαν υποχρέωση δήλωσης ΦΥΠΙΑ Κανονικά, μία φορά τριετία ε, ε, κάθε έμπορος ε, θα είχε μια επίσκεψη εφοριακού ανεξαρτήτως μεγέθους. Τώρα αυτό έχει γίνει μια φορά στα 300 χρόνια. Έχουν εξαφανιστεί οι εξωτερικοί έλεγχοι και θα πρέπει να επανέλθουν γιατί έχουν πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα. γιατί έχουμε καθημερινά ε, απάτη στην αγορά. Ευχαριστούμε. Έχουμε πάλι χρόνο για το ΕΛΚΟ, κύριος Φαντακαντέλα. Ζητώ συγγνώμη που θα σας ξανακουράσω με μια ερώτηση στα Ολλανδικά και θα πρέπει να βάλετε τα ακουστικά σας. Κύριε Αλοψωτήρη, έχω συγκεκριμένη ερώτηση για την πρωτοβουλία Eurofisk και σας ευχαριστώ καταρχάς για όσα μας είπατε. Είναι καλή πρωτοβουλία ε, και χρήσιμη. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι όλα τα... μπορεί να είναι όλα τα κράτη-μέλη μέρη στο Eurofisk, αλλά επειδή είναι θελοντική συμμετοχή ε, δεν έχει μεγάλη αποτελεσματικότητα και υπάρχει και μικρή διαφάνεια για το ποιο κράτος μέλος συμβάλλει με ποιο τρόπο. Θα μπορούσατε να μας δώσετε μια εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη συνεισφέρουν, ποια συνεισφέρουν τα περισσότερα, ποια τα λιγότερα, ποια ε, είναι εκείνα που είναι πιο δραστήρια και ποια λιγότερα. Είναι της μόδας τώρα το naming and shaming, οπότε μην διστάσετε. Και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε για να λειτουργεί καλύτερα το δίκτυο. Θα αλλάξει με το νέο σύστημα τίποτα στη λειτουργία του Eurofisk. Yes, Mrs. Κυρία Όλαφ Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των κρατών μελών, είναι λογικό και σωστό τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν. και όταν μιλάμε για τους κοινού τομεί εργασία, είναι υποχρεωμένα τα κράτη-μέλη να ανταλλάσσουν και πληροφορίες βάσει του τι συμφώνησαν τα μέλη της ομάδας εργασίας για αυτό το συγκεκριμένο τομέα. Είναι μέρος λοιπόν της διαδικασίας των κρατών μελών ε, να αποφασίσουν τι πληροφορίε θα ανταλλάσσουν. Η συνεισφορά στο δίκτυο εξαρτάται από την κλίμακα της απάτης στο κάθε μέλος. Και στα 28 το επίπεδο της απάτης και των εταιριών που το διαπράττουν είναι πολύ διαφορετικό. Αυτό σημαίνει ότι σε μεγάλες χώρες, με πολλές εταιρείες, που υπάρχει και πολλή απάτη, προφανώς δίνουν περισσότερες πληροφορίες για συναλλαγές, υπόπτες συναλλαγές, προς το δίκτυο. Πάντως είναι σημαντικό όλες οι εθνικές αρχές να εντοπίζουν τις εταιρείες που διαπράττουν απάτη σε εθνικό επίπεδο και μετά να τροφοδοτούν αναλόγως στο σύστημα. Η δεύτερη ερώτηση Α, ναι, πώς να γίνει υποχρεωτικό. Δεν είναι υποχρεωτικό, όπως είπαμε, να συμμετέχει κανείς στο Eurofisk και δεν είναι και υποχρεωτικό να ανταλλάσσονται αυτέ τις πληροφορίε. Οπότε νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει υποχρεωτικό για τα κατημέλη να συμμετέχουν. Είναι εθνική η απόφαση. Ναι, αλλά ας φανταστούμε ότι θα μπορούσαμε. Μήπως θα ήταν πιο αποτελεσματικό από ό,τι είναι σήμερα το σύστημα. Μα είναι τελείως θεωρητική η ερώτησή σας. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται, γιατί και τα 28 κρατη συμμετέχουν στο δίκτυο και σχεδόν όλα τα κρατη σχεδόν όλα, συμμετέχουν σε όλου του τομεί εργασία. Οπότε τα κράτη-μέλη, ακόμη και θελοντικά, δίνουν, δίνουν πολύ ε, από τους πόρους τους και από τις πληροφορίες τους. Έχουν καταλάβει ότι έχει κάποιο αποτέλεσμα αν ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο. Σε κάποια φάση όλα τα κράτη-μέλη μπορούν να υποστούν σοβαρές απώλειες και κανείς δεν ξέρει ποτέ ποιο θα είναι το επόμενο κράτος που θα είναι στόχος. Ευχαριστούμε πολύ η ε, αντιπρόεδρος μας, η ε, κυρία Γκόμες. Να σχολιάσω αυτό που είπε ο κύριος Μέρφυ. Ναι, η ψηφιοποίηση του πορτογαλικού συστήματος ήταν χρήσιμη. Αλλά για τις μικρές επιχειρήσεις και για τα άτομα όπως ένας κομμωτής ή ένας που έχει συνεργείο αλλά επειδή δεν έχει επαρκείς πόρους ε, η εφορία, δεν ελέγχει τις μεγάλες επιχειρήσεις και τους ε, πλουσίους. Και το λαχείο ε, επίσης ε, καταργήθηκε γιατί ήταν απαράδεκτο. Ήταν ένα κόλπο για να πουλάνε γερμανικά αυτοκίνητα. Ναι, έχει βελτιωθεί το σύστημα. και έχει επηρεάσει τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Έχω καταλάβει τώρα πληρώνουν φόρους. Μια ερώτηση προς την Κομισιόν. Εφόσον ξέρετε τι παίζετε για τους ίδιους πόρους της Ένωσης και ενώ τώρα συζητάμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για την επόμενη ετία, Και επειδή είναι σαφές όπως ακούσαμε στην προηγούμενη συζήτηση ότι οι απώλειες ΦΠΑ λόγω απάτης χρηματοδοτούν την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα. Πώς είναι δυνατόν να μην είναι η πρώτη προτεραιότητα των κρατών μελών αλλά και της Επιτροπής της ίδιας. Πώς είναι δυνατόν να θέσουν τα κράτη-μέλη, να θέσει η Επιτροπή τα κράτη-μέλη ενώπιον ε, των ευθυνών τους. Γιατί δεν ξέρουμε ποιες χώρες αντιπαρατίθενται. Αν δεν μπορείτε να μας πείτε τώρα, να μας πείτε αργότερα. Ποιες χώρες είναι κατά για να τις θέσουμε εμείς ενώπιον των ευθυνών τους. Και μία ερώτηση προς όλους. Λόγω των επιπτώσεων των κρυπτονομισμάτων. Για κάθε είδους ε, συναλλαγές Ακόμη και κάποια κράτη-μέλη θέλουν να είναι κέντρα κρυπτονομισμάτων. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις λοιπόν αυτής της χρήσης των κρυπτονομισμάτων. Ο πρόεδρος, ναι, ξέρει η Κομισιόν θα μας τις πει όμως τις χώρες αυτές. Για να δούμε, ορίστε. χαίρομαι που δεν μου ζητείτε να αποκαλύψω το κατάλογο. Βεβαίως το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο πρόεδρος Γιούνκερ ε, έδωσε εντολή στον Επίτροπο Μοσκοβισή και ήταν ξεκάθαρο ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να έχουμε μια σαφή πρωτοβουλία για μια πολιτική καταπολέμηση απάτης ΦΠΑ. Αλλά και γενικά τα φορολογικά, φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή είναι προτεραιότητα ύψιστη ε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Επίτροπο Μοσκοβισή που ήταν ιδιαίτερα δραστήριος και δημόσια με επισκέψεις στα κρατη αλλά όχι μόνο δημόσια. Πιέζει και τα κρατη να κάνουν προσπάθειες έτσι ώστε να καταπολεμούν ε, τις ε, απάτες στα φορολογικά, ιδιαίτερα στο ΦΠΑ. Βεβαίως έχουμε προτάσεις και πρωτοβουλίες και φέρουμε τη συζήτηση ε, στο τραπέζι του Συμβουλίου για να συζητήσει τις προτάσεις. Καμιά φορά, πηγαίνει, μάλλον σε τακτά χρονικά διαστήματα, φτάνουν και στο Υπουργικό Συμβούλιο και ακούμε και τις θέσεις των διαφόρων κρατών μελών στο ΕΚΟΦΗΝ κτλ. Έχουμε προτάσεις, έχουμε και συνοδευτικά μέτρα στη συνεδριάση με τους επικεφαλείς των εφοριών για να μπορούν να συνεργάζονται καλύτερα και να αξιοποιούν καλύτερα την εσωτερική αγορά γιατί αυτό είναι ένας από τους στόχους και να υπάρχει και ε, ίσπραξη των φορολογικών εσόδων που δικαιούνται και να συνεισφέρει και ο κρατικός προπολογισμό στον Ευρωπαϊκό. Τι γίνεται με τα κράτη-μέλη που δεν εφαρμόζουν σωστά την νομοθεσία. Θα πρέπει να αναλυφθεί δράση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ε, καμιά φορά έχουν ε, κακή ερμηνεία της νομοθεσίας ή ακόμα και έλλειψη πόρων ή δεν είναι σωστές οι διαδικασίες και ε, όσα εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να συμμορφώνονται οι πολίτες. Δηλαδή έχουμε τριπλή δράση. Έχουμε σε πολιτικό επίπεδο ε, με σαφή μηνύματα από τα θεσμικά όργανα και εσείς ακούτε συχνά. Ε, το δεύτερο είναι η νομοθετική δράση και η τρίτη επιβολή του νόμου. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι σε όλα τα κράτη-μέλη με τον ίδιο τρόπο εφαρμόζεται ο νόμος. Α, και ένα τέταρτο που είναι οι βοήθειες στις φορολογικές αρχές για να έρχονται σε επαφή, να συνεργάζονται ε, με το Eurofisk που είναι ένα δίκτυο, αλλά υπάρχουν και άτυπες συζητήσεις και επαφέ που έχουν μεταξύ τους έτσι ώστε να βρουν κοινέ λύσει για τα κοινά προβλήματα, γιατί είναι κοινά τα προβλήματα. Κύριε ένα σύντομο σχόλιο για την πρώτη σας παρατήρηση, διότι όντω στον ε, τωρινό μου ρόλο και με τον τωρινό μου ιδιότητα ως καθηγητή που στο Πανεπιστήμιο ασχολούμαι με τα θέματα της φορολογίας είμαι εντελώ απομονωμένος και ε, ακόμη και το εγχείρημα να συνεργαστώ με άλλους ε, στα πλαίσια του ακαδημαϊκού χώρου είναι πολύ ε, απομονωμένο το να δημοσιεύονται άρθρα για τη φορολογία από μικροοικονομική σκοπιά ε, σε οποιασδήποτε επιστημονικές εφημερίδες είναι κάτι, το να κάνει κανείς έρευνα μπορεί να γίνει αλλά ως προς την επικοινωνία οι μακροοικονομολόγοι ούτε που ασχολούνται με αυτές τις θεωρίες είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να προβληθούν τα φορολογικά θέματα, ελάχιστα ενδιαφέρονται. Αυτή λοιπόν η αδιαφορία είναι τόσο εξαπλωμένη γιατί η μόνη που ε, έχει η μόνη που ενθουσιάζεται με τα φορολογικά θέματα είναι η γυναίκα μου που έχει διαγνωστεί και με συγκεκριμένη πάθηση. Ε, υπάρχει βεβαίως το κρυπτονόμισμα που είναι το αντίστοιχο του φορολογικού παραδείσου και πρέπει λίγο να το αντιμετωπίσουμε. Διάλλως ε, υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Πρέπει κάποια πράγματα να αποκαλύπτονται αν οι συναλλαγήσουν σε κρυπτονόμισμα και δεν υπάρχουν ε, στοιχεία για, τα στοιχ... για, την... Ε, για τις λεπτομέρειες της συναλλαγή και δεν μπορούν να κοινοποιηθούν στη φορολογική αρχή, τότε δεν μπορούν να εφαρμοστούν ε, οι κανόνες και οι διατάξει του νόμου με τον οποίο η νομοθεσία του νόμου και τη νομοθεσίας του κράτους εντό του οποίου γίνεται αυτή η συναλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να ισχύει το σύστημα επιβολής του νόμου για τα φορολογικά. Πρέπει λοιπόν να είμαστε τόσο ξεκάθαροι με, τους, ε, με τα κράτη που επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Ότι δεν θα έχετε προσβάσει στο νομικό σύστημα και η διαφάνεια αυτή δεν σα επιτρέπει να πάρετε πίσω το εισόδημα που σα αναλογεί από το ΦΠΑ. Πρόεδρο, δεν βλέπω κάποιο άλλο να ζητά το λόγο. Σε αυτή την περίπτωση να ζητήσω από τον συνεισηγητή μα, τον κύριο Νίντερμαϊ, να μα πει αν θέλει το λόγο για καταληκτήριε παρατηρήσει. Όχι. Να ευχαριστήσω πολύ λοιπόν τους φιλοξενούμενούς μας για τις εισηγήσεις τους, τις παρατηρήσεις τους, όσα μας είπαν για την κυκλική απάτη και το φόρο ΦΠΑ, την απάτη του φόρου ΦΠΑ. Είδαμε τι προοπτικές υπάρχουν για το μέλλον Σίγουρα δεν θα έχουμε ολοκληρώσει πρωτού υπάρξει ένα οριστικό ε, σύστημα ΦΠΑ που να εξετάζεται ως πρόταση από το Συμβούλιο. Όμως λόγω, του, όμως λόγω του όγκου και του ποσού των χρηματικών ποσών που έχουν να κάνουν με την απάτη ΦΠΑ δεν είναι πιθανό παρόλο που δεν είναι να συμβεί άτομο, να συμβεί άμεσα, είναι ένα από τα μείζωνα ζητήματα που θα θέσει η Επιτροπή μα και στα πλαίσια του σκόρμπορ, του βαθμολογίου. Ελπίζουμε ότι θα σκεφτεί περισσότερη πίεση στι εθνικέ κυβερνήσει να βρουν λύσει για το κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τρόπο αποτελεσματικό. Επόμενη συνεδρίαση τη Επιτροπή αυτή τον Σεπτέμβριο. Εν τω μεταξύ θα έχουμε και αποστολή της Επιτροπής στην Washington θα συναντήσουμε τον ε, Υπουργό Οικονομικών, ε, την εκπροσώπους της Φίνσεν, θα πάμε στο Κογκρέσο. Αυτό είναι το πρόγραμμα για τις ερχόμενες εβδομάδες. Το σημείο μου λέει να σας πω καλές διακοπές, αλλά δεν θα ήθελα να ξεχάσετε ότι την επόμενη εβδομάδα πάμε και στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο. Θα πάμε λοιπόν και στο Στρασβούργο και πάλι ευχαριστώ πολύ τους προσκεκλημένους μας. Ε, κυρίως τη λήξη της